Για να αρχίσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε ως προσωρινός πρόεδρος και πραγματικά προσωρινός κηρύσω την έναρξη της συνεδρίας. Έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες. Σύμφωνα το φως του Προεδρείου του Κοινοβουλίου. Στόχο τη συνεδρίαση είναι η σύστηση σε σώμα του Προεδρείου τη Υποεπιτροπή μέσω τη εκλογή Προέδρου και τεσσάρων αντιπροέδρων. Σύμφωνα με το άρθρο 2.13 του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου μα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα εκλογή Προέδρου και κατόπιν ε, αντιπροέδρων. Οι αναπληρωτέ που συμμετέχουν είναι οι εξή. Μα ενημέρωσαν ότι η Σίλβια Σαντώνη του IND θα, θα αντικαταστήσει τον ε, Πατρίκ Μπέρκ. Έχουμε απαρτία, άρα οι ψηφοφορίε είναι έγκυρε, τουλάχιστον 8, το 1 τέταρτο, δηλαδή των μελών, το επιβεβαίωσε η γραμματεία. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι τους άλλους, όπως διαπιστώνω στην αίθουσα. Δεν είναι και πολύ απαιτητικό ο εσωτερικό κανονισμό για την απαρτία. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι οι υποψηφιότητε μπορούν να υποβληθούν είτε από μια πολιτική ομάδα είτε από τουλάχιστον δύο συναδέλφου, ένα εικοστό δηλαδή των μελών τη Επιτροπή μα. Οι υποψηφιότητε πρέπει να υποβληθούν με τη συμφωνία των υποψηφίων. Οι υποψήφοι πρέπει να είναι τακτικά μέλη της Επιτροπής και πρέπει να έχουν ε, συμπληρώσει την ε, δήλωση οικονομικών συμφερόντων και κατάλληλη συμπεριφορά. Η σύνθεση του Προεδρείου πρέπει να αντικατοπτρίζει την ε, ποικιλότητα του Κοινοβουλίου δεν μπορεί να είναι μόνο άντρε ή γυναίκε και όλοι οι αντιπρόεδροι δεν μπορεί να προέρχονται από το ίδιο κράτο μέλο με βάση το άρθρο 2.13 του εσωτερικού κανονισμού. Όλα τα τακτικά και πραγματικά μέλη που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία πρέπει να έχουν την ε, κάρτα του εάν γίνουν ηλεκτρονικέ ή μυστικέ ψηφοφορίε. Καλό τι πολιτικέ ομάδε να προτείνουν υποψηφιότητε για την Προεδρία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από πλευρά των σοσιαλιστών προτείνω την κυρία Μαρία Αρενά για Προεδρία. Μάλιστα, είναι τακτικό μέλος της Υποεπιτροπής και της ΑΦΕΤ και έχει συμπληρώσει και τις δηλώσεις. Εντάξει, έτσι, έτσι δεν είναι. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Και δέχεστε και την υποψηφιότητα. Τι δέχεστε. Πολύ ωραία. Οπότε η εκλογή της ε, Μαρία Αρενά μπορεί να γίνει διαβοής. Αν υπάρξει βοή, είστε πρόεδρος. Ευχαριστώ που στήριξατε κυρία ε, Αρενά με ενθουσιώδης ενθουσιώδε χειροκρότημα. Παρακαλώ, ελάτε. Merci, merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη που μου χορηγείτε μέσω αυτής της εκλογής μου δια βοή. Ξέρω ότι ευθύνη έχει η πρόεδρος μια υποεπιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσοι με γνωρίζουν, ξέρουν ότι θα αγωνιστώ, θα κάνω ό,τι μπορώ για να προασπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην Ευρώπη για την τμήμα των συνθηκών, των αξιών μας, του γονιδιώματός μας και σε όλες τις εξωτερικές σχέσεις που έχουμε. Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα είναι φυσικά κύριο μέλημά μας. Χάρη στην δική σας εργασία, ανεξαρτήτως ε, πολιτικής τοποθέτησης, βεβαίω ενδιαφέρεστε να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον Σάρλ για την μεταβατική του Προεδρία, τη σύντομη. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα και είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε πολύ κατά την προηγούμενη θητεία. Ευχαριστώ πολύ για όσα ήδη έκανες μέχρι τώρα. Οπότε, η διάταξη. Θα εκλέξουμε τώρα τους αντιπρόεδρους. Διαδικαστικά. Έχουμε φυσικά απαρτία, άρα η ψηφοφορία είναι έγκυρη και οι επόμενε θα είναι. Παρακαλώ τις πολιτικές ομάδες να με ενημερώσουν για υποψηφιότητε για την πρώτη αντιπροεδρία. Παρακαλώ. Εξ ονόματο ομάδα Renew Europe θα ήθελα να προτείνω την κυρία Φονβίζερ για πρώτη ε, αντιπρόεδρο. Σας ευχαριστώ. Είναι μέλος της Υποεπιτροπής και της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Έχει συμπληρώσει την ε, δήλωση για τα οικονομικά συμφέροντα και για τον κώδικα δεοντολογίας. Αποδέχεστε την πρόταση. Μάλιστα, ευχαριστώ. Καθότι έχουμε μία και μόνη υποψήφιο ως πρώτη αντιπρόεδρο, σας προτείνω διαβοήσει να εκλέξουμε. Σας ευχαριστώ. Αν θέλετε να έρθετε κι εσείς εδώ στο βήμα. Λοιπόν, πάμε στην, ε, στο δεύτερο αντιπρόεδρο. Έχουμε απαρτία. Σας ζητώ να παρουσιάσετε την υποψηφιότητα, παρακαλώ. Ε, πρόεδρε, θα ήθελα να προτείνω ως δεύτερη αντιπρόεδρο την κυρία Χάνα Νόημα από τους Πρασίνους. Σας ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Είναι πλήρες μέλος της Υποεπιτροπής και επίσης μέλος της ΑΦΕΤ. Έχει συμπληρώσει τα σχετικά έγγραφα του κώδικα και των οικονομικών συμφερόντων. Αποδέχεστε την υποσιότητα. Ναι, πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Σας ζητώ να εκλέξουμε διαβοήση εφόσον δεν έχουμε έτοιμα μυστικής ψήφου. Σας ευχαριστώ. Αν θέλετε, ελάτε κι εσείς εδώ στο βήμα. Nous allons maintenant passer à la troisième. Τρίτος αντιπρόεδρος τώρα, ίδια διαδικασία. Παρακαλώ την ομάδα να παρουσιάσει την ε, υποψηφιότητα για τον τρίτο αντιπρόεδρο. Παρακαλώ. Να σας συγχαρώ, Πρόεδρε, για την εκλογή σας και εκ μέρους του ΕΛΚ να προτείνω την Καρολίνα Ετστάκλερ για τρίτη αντιπρόεδρο. Ναι, επαναλάβω ότι είναι μόνιμο μέλος της Υποεπιτροπή και μέλος της Επιτροπής ΑΦΕΤ, έχει συμπληρώσει τις σχετικέ δηλώσεις που απαιτούνται ή κυρία αποδέχεται την ε, υποψηφιότητα. Μάλιστα, Πρόεδρε, σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Εφόσον έχουμε μία και μόνη υποψήφιο, παρακαλώ να σφίσουμε διαβοή. Να εκλέξουμε. Bienvenue, je vous propose de venir nous rejoindre. Ελάτε κι εσείς εδώ στο βήμα. Λοιπόν, θα σημειώσατε ότι έχουμε μέχρι εδώ προεδρείο αποκλειστικά με γυναίκες και ο κανονισμός μας επιβάλλει να υπάρχει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος του άλλου φίλου. Έχουμε λοιπόν την υποψιότητα του τέταρτου αντιπροέδρου, παρακαλώ, τις ομάδες ο κ. Κιούρενς ε, παρότι το Προεδρείο θα μπορούσε να είναι μόνο γυναίκες ήθελα να πω ότι εμείς εδώ στο Renew δεν ενοχλούμαστε καθόλου από αυτό. Έχετε ε, κάποιο, έχετε, θέλετε το λόγο επί της διαδικασίας με μικρόφωνο παρακαλούμε. Κοιτάξτε, οι κανόνες λένε ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία των φίλων. ισορροπία λέει, όχι απλώς και μόνο ένας. Εγώ σε τρεις επιτροπές σήμερα ήμουν παρόν και ακύρωσαν, ανέβαλαν την ψηφοφορία. Γιατί δεν είχαν εκπρόσωπο. Ένας και μόνο άνδρας δεν είναι η ισορροπία των φίλων. Ε, νομίζω ότι η διάσκεψη των Πρόεδρων μπορεί να έχει αντίθετη γνώμη, Πρόεδρε. Η πρόεδρος λέει οι κανόνες είναι σαφείς. Θα έχουμε τώρα την πρώτη υποψιότητα για τον τέταρτο αντιπρόεδρο σας παρακαλώ. Ιζαμπέλ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, να σα συγχαρώ για την εκλογή σα. και να υποβάλλω την υποψηφιότητα του Ράφαελ Γκλούξμαν ως ε, τέταρτου αντιπροέδρου. Ναι, νομίζω είναι άνδρας, λέει η πρόεδρος. Λέω νομίζω, παραλαμβάνει η πρόεδρος. Τακτικό μέλος της υποεπιτροπής και μέλος της Επιτροπής ΑΦΕΤ, έχει δηλώσει τα απαραίτητα έγγραφα, όπως και οι προηγούμενοι υποψήφοι, αποδέχεστε την υποψηφιότητα, αποδέχομαι με τα χαράς Πρόεδρε. Σας προτείνω διαβοής, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ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 για τη συγκρότηση του Προεδρείου. Το επόμενο σημείο είναι η γλωσσική κάλυψη και το ημερολόγιο για το 19 για, το, για τη γλωσσική κάλυψη της υποεπιτροπής. Σύμφωνα με την συγκρότηση και τους κανόνες τους εφαρμοστέους θα υπάρχουν 13 γλώσσες γερμανικά, γερμανικά αγγλικά, γαλλικά φιλανδικά, ελληνικά, ουγγρικά, ιταλικά, ολλανδικά, πορτογαλικά, ρουμανικά και σουηδικά. Αυτό κατά τις επίσημες συνεδριάσεις της υποεπιτροπής, συνεχίζει η πρόεδρος. Δεν έχουμε σχόλια από αυτού. Ωραία. Για τις συνεδριάσεις θα λάβατε το ημερολόγιο για το 19 δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν δεν έχουμε άλλα σχόλια, θεωρώ ότι το έχουμε εγκρίνει. Αν δεν έχουμε αντίρρηση. Ωραία. Το τέταρτο σημείο είναι η πρώτη συνεδρίαση του Διευρυμένου Προεδρίου για την Δευτέρα 15 Ιουλίου μεταξύ 7 και 8 το βράδυ. Η Γραμματεία θα εμπεβαιώσει και το της ώρας και το της αιθούσης το συντομά των δυνατών. Δεν έχω άλλα σημεία για σήμερα, επομένως ολοκληρώνουμε για σήμερα. Ευχαριστώ όλους.